Φίλοι μου, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Έχουμε καθυστερήσει και μερικά λεπτάκια, αλλά έχουμε ενώπιόν μας ε, τρεις ώρες ψηφοφορίας. Four minutes Ας μην καθυστερήσουμε λοιπόν πιο πολύ. Τρεις ώρες έχουμε μπροστά μας λίγο πολύ και να ξεκινήσουμε με μία δοκιμαστική ψηφοφορία, παρακαλώ. Δοκιμαστική ψηφοφορία, παρακαλώ, βάλτε τις κάρτες στα μηχανήματα. Έναρξη της ψηφοφορίας. Πέρας. Πολύ ωραία. Όλα λειτουργούν τέλεια. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε ευθύς εξ αρχής δύο εκθέσεις. Με 4.500 τροπολογίες από κοινού. Οι εισηγητές. Η πρώτη είναι η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου έρευνα και καινοτομία Ορίζον Ευρώπη. Νταν Νίκα, ο εισηγητή. Η δεύτερη τα έκθεση θα είναι εφαρμοστική. Να ξεκινήσουμε με την πρώτη, με τον ορίζοντα Ευρώπη. Νταν Νίκα. Συμβιβασμός 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές αποδεκτό. Συμβαστικό 2. Συμβασμό 2. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβασμό 3. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 6α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Υπέρ περιμένω, λέει ο πρόεδρο. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ Διορθώνει ο πρόεδρο. Πήδηξα μία σελίδα. 16 συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ.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 κατά αποχές έγκρινεται. 29 υπέρ, κατά αποχές έγκρινεται. Συμβαστική 30 υπέρ, κατά αποχές έγκρινεται. Συμβαστική 31 υπέρ, κατά αποχές έγκρινεται. 32 υπέρ, κατά αποχές έγκρινεται. 33. Έλεγχος. Για την συμβαστική 32 ζητείται έλεγχος. Έναρξη ψηφοφορίας. Από τους σοσιαλδημοκράτες περισσεύει ένας. Ένας είναι υπεράριθμος. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ για το διάλειμμα. Η 33, υπέρ. Κατά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 κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Α3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Α4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Α5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. R1 υπέρ κατά αποχές έγκρινε. Αρ2 υπέρ κατά αποχές έγκρινε. Αρ2α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. έγκρινε. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. έγκρινε. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αρ5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. R5α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. R6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. R7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. R8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. R8α υπέρ κατά αποχές αποδεκτή. R8β ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. R 8C ε, υπέρ κατά αποχές R 8D ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται R 9 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται R 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται R 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται R12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνεται. R12α υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. R13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. R14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. R15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. R16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. R17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. R18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. R19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. R20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. R21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. R22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. R 23 υπέρ. Κατά. Αποχές Αρ R24 υπέρ. Κατά. Αποχές Αρ R25 υπέρ. Κατά. Αποχές Αρ R26 υπέρ. Κατά. Αποχές Αρ R26 β υπέρ. Κατά. Αποχές Αρ R27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. R28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. R29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. R31 unblock υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. R39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. R40 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. R41 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. R43 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. R45 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. R47 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. R48 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. R49 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται R50 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται R51 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται R52 unblock υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για το σχέδιο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Με ονομαστική κλίση ασφαλώς. Έναρξη της ψηφοφορίας. Ένας υπεραριθμός από το ΕΛΚ, δύο από το ΕΛΚ και από τους σοσιαλδημοκράτες. Δύο από το ΕΛΚ, ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς, δυστυχώς. Και άλλος ένας. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μάλιστα. τη ψηφοφορία τώρα. Πολύ καλά αποτελέσματα και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ο εισηγητής θέλει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Κιώδης ε, για την σκληρή τους εργασία τους δύο αυτούς μήνες, επίσης τους βοηθούς, τους εμπειρογνώμονες των πολιτικών ομάδων. Δεν θα σας πω καν πόσες συναντήσεις ε, σκιωδών είχαμε. Το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό και ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας βοήθησε ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε το Γενικό Διευθυντή και όλους σας. Είναι εξαιρετική έκθεση, είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και νομίζω ότι πρέπει να συγχαρούμε τους πάντες για αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ωραία, σας ευχαριστώ. Τώρα αγαπητοί φίλοι θα ψηφίσουμε τη δίδυμη έκθεση της προηγούμενης γιατί ε, είναι ομοειδείς αυτές οι εκθέσεις και γεννήθηκαν την ίδια στιγμή. Ναι, κάτι θέλετε να πείτε, έχετε το λόγο. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος είναι κατά της ψηφοφορίας unblock, γιατί έτσι θα κερδίσουμε πολύ χρόνο, αν δεν αντιτίθεται δηλαδή κανείς. Άρα περνάμε στην τελική ψηφοφορία, λέει κάποιος ε, χαριτολογώντας. Okay, so is my, is my question. Συμφωνείτε για την ψηφοφορία μπλοκ. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Άρα, ο κύριος Κρίστιαν Έλλερ είναι ο εισηγητής και θα ήθελε να αποφασίσουμε για το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την υλοποίηση του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη, πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας. Ο κύριος Κρίστιαν Έλερ είναι ο εισηγητής και αρχίζουμε με την ψηφοφορία. Συμβαστική 1. Υπέρ. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Ε, Αγαπητοί φίλοι, κατανοώ ότι είσαστε έτοιμοι να ψηφίσετε για δύο λεπτά και να μην τα υπερβούμε. Ωραία. Εγώ θα τα καταφέρω. Άμα θέλετε και για μισή ώρα μπορώ να σας μιλάω, να σας λέω υπέρ κατά Ωραία, με ονομαστική κλίση. Λοιπόν, αν ψηφίσουμε ολόκληρη την έκθεση unblock, Uh, Δύο ψηφοφορίες θα έχουμε. Μία για όλες τις συμβαστικές unblock και τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Ωραία. Δεν το κατανόησα γιατί είναι τόσο εύκολο που κατέστη δύσκολο. Δυσνόητο. Λοιπόν, unblock ψηφίζουμε όλες τις συμβαστικές τροπολογίες. και μετά θα έχουμε ονομαστική κλίση για το σύνολο της έκθεσης. Λοιπόν, αρχίζουμε φίλοι. Ονομαστική κλίση, μπορείτε να το δεχτείτε αυτό, αυτή τη διαδικασία. Άρχεται η ψηφοφορία επί της διαδικασίας. One EPP too many. Ένας υπεράριθμος από το ΕΛΚ. Κρίστιαν, εντάξει, εντάξει. Εγώ έβγαλα τη δική μου ψήφο. Πέρας. Όλοι τάσσονται υπέρ. Τώρα, Κρίστιαν, βάζω την κάρτα μου και έχουμε ονομαστική για το σύνολο της έκθεσης όπως έχει τροποποιηθεί. Τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση, η οποία και άρχεται. Okay. No. Ένας υπεράριθμος πάλι από το ΕΛΚ. And close the Πέρας. Εξαιρετικό αποτέλεσμα. 61 Συγχαρητήρια προς το συνάδελφο. Και άρα θα ψηφίζουμε για δύο ώρες, όχι τρεις. Ο κύριος Έλερ έχει το λόγο. Απλώς ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν το προσωπικό, τη γραμματεία, και όλους τους συμβούλους που εργάστηκαν, γιατί γράφουμε ιστορία τώρα, μην το ξεχνάτε. Είναι το τρίτο ερευνητικό πρόγραμμα και δεν πιστεύουμε ότι δεν θα το ε, καταφέρναμε να ψηφίσουμε όλες τις ε, συμβαστικές. Στέλνουμε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στο Συμβούλιο ότι αρχίζουμε τις διαπραγματεύσεις και θέλουμε αποτέλεσμα πριν από το τέλος της θητείας γιατί το χρειάζεται η Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε συνάδελφοι. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Ε, κύριοι Έλερ και Νίκα. Και θα ήθελα να συγχαρώ και όλους τους σκιώδεις. Ένα θερμό ευχαριστώ. Δέκα συνάδελφοι εργάστηκαν ε, πολύ καλά. Τώρα, θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 21-27. Η Αγγέλικα Μλίναρ είναι η συγγήτρια και αρχίζουμε άμεσα. Καλτ 27 υπέρ. Κατά αποχές αποδεκτή. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές αποδεκτή. 18 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 19 υπέρ κατά αποχές αποδεκτή. Κάλτ 29 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 20 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Ήμκο 46 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Τι θέλετε. Θέλετε να ελέγξουμε. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε λοιπόν ΙΜΚΟ 46. ΙΜΚΟ 46. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Με συγχωρείτε. Κάνε λάθος. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Παρακαλώ να σηκώνετε το χέρι γιατί δεν σας βλέπω και δεν μπορώ να υπολογίσω. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συνάδελφοι εξ αριστερών να σηκώνετε το χέρι. Δηλαδή να είναι ορατό. Συμβαστική 7. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. unblock. Μπλοκ 1 μάλλον. Όλες οι τροπολογίες για τον προϋπολογισμό. Υπέρ, κατά, αποχές δεκτές. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Budget 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 294 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 52 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 53 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές ε, δεκτή 63 υπέρ. Κατά αποχές ΙΜΚΟ 80 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε την ΙΜΚΟ 80. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένας πάλι υπεράριθμος από το ΕΛΚ. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή 70 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή 338 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 347 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ίμκο 88 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 348 υπέρ, κατά. Ας ελέγξουμε καλύτερα. 348 άρχεται η ψηφοφορία και πέρας. Απορρίπτεται. Καλτ 57 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή τραν 56 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή τραν 57 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή τραν 58 υπέρ. Κατά αποχές αποδεκτή τραν 59 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή Θέλετε να ελέγξουμε. Τραν 59. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Και εγκρίνεται. Ε, κάλτε 61 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Κάλτε 62 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Κάλτε 63 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Τραν 60 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Καλτ 64 υπέρ, κατά. Ας ελέγξουμε καλύτερα. Καλτ 64, πέρας. Αποδεκτή. Ήμκο 89. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε την Ήμκο 89. Πέρας. Δεκτή. Ήμκο 90. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Καλτ 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Κάλτε 67 υπέρ κατά. Ας ελέγξουμε. Καλτ 67. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Και εγκρίνεται. Καλτ 68. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε, ας ελέγξουμε καλύτερα. Καλτ 68. Πέρας. Δεκτή. Ήμκο 91 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Αμπλοκ 75, 76, 77, 78. Υπέρ κατά αποχές αποδεκτές 92 ΙΜΚΟ υπέρ κατά αποχές αποδεκτή 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή όλες οι γιούρι αμπλοκ υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 61 υπέρ κατά Ας ελέγξουμε την τραν 61. 61. Τραν 61 πέρας. Αποδεκτή ΙΜΚΟ 93 υπέρ. Κατά. Αποχές αποδεκτή. Ε, 94 υπέρ. Κατά αποχές αποδεκτή. 352 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε 352 πέρας απορρίπτεται 353 υπέρ κατά ας ελέγξουμε πέρας απορρίπτεται αυτή τη φορά 354 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Κάλτε 72 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Κάλτε 73 υπέρ, κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Ήμκο 96 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Κάλτε 74 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 356 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 97 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Ήμκο 98 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Ήμκο 99 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 357 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 100 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 358 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται τραν 62 υπέρ κατά αποχές δεκτή 359 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε καλύτερα πέρας ένας υπεράριθμος από το ΕΛΚ τώρα κλείνω και απορρίπτεται Transport 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 360 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε την 360 πέρας και απορρίπτεται. Κάλτε 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Κάλτε 77 υπέρ, κατά. Ας ελέγξουμε. Καλτ 77. Ελέγχουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Καλτ 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 361 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται κάλτε 75 υπέρ κατά αποχές αποδεκτή 362 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ΙΜΚΟ 104 υπέρ κατά αποχές δεκτή 363 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Κάλτε 79 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Κάλτε 80 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 364 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 365 υπέρ. 364 να ελέγξουμε θέλετε εντάξει. Έλεγχος. Rejected. Rejected. 365 in favor. 365 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν δεν σηκώνετε τα χέρια δεν αποφασίζουμε. Ας ελέγξουμε, παρακαλώ. 365 ελέγχουμε. I close the vote. Πέρας. Αποδεκτή. Ήμκο 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ήμκο 102. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ήμκο 103 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Κάλτο 81 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Ήμκο 105 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Ήμκο 106 υπέρ κατά αποχές δεκτή. ΙΜΚΟ 107 υπέρ. Κατά αποχές. Ας ελέγξουμε, ας ελέγξουμε. 107 ήμκο ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρασε. Και απορρίπτεται. Κάλτο 82 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Κάλτ 83 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Καλ... Α, 80, 80 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Κάλτ 1 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Λίμπε 1 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Ήμκο 1 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Καλτ 2 υπέρ, κατά, Ας ελέγξουμε την Καλτ 2. Πέρας. Απορρίπτεται. ΙΜΚΟ 2 υπέρ. Κατά. Αποχές αποδεκτή. ΛΥΜΠΕ 2 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 81 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε την 81. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή 83 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε την 83. 83 ελέγχουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Καλτ 3 υπέρ κατά αποχές αποδεκτή λίμπε 3 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 84 υπέρ, κατά ας ελέγξουμε 84 ελέγχουμε πέρας απορρίπτεται ΙΜΚΟ 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή λίμπε 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 86 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή συμβαστική 16 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 33 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή λίμπε 5 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 91 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 93 υπέρ. Κατά αποχές ας ελέγξουμε την 93 έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ήμκο 5 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 298 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε 98 98 τι να κάνω Πατρίτσια κανένας δεν σκονεί το χέρι του πέρας 55 προς 3. Αγαπητοί φίλοι, να σηκώνετε το χέρι σας για να βλέπω. Πρέπει να κάνετε μια προσπάθεια. Καλτέξι, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 6 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή τραν 6 υπέρ. Κατά. Αποχές ας ελέγξουμε την τραν 6 έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. Ήμκο 7 υπέρ. Κατά. Αποχές θα πρέπει να ελέγξουμε. Ήμκο 7. Έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται με μικρή διαφορά. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ήμκο 9 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Αμπλόκ τώρα ψηφίζουμε την 109, ΙΜΚΟ 11, ΤΡΑΝ 7, αμπλόκ, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές, 112 υπέρ κατά αποχές δεκτή 115 υπέρ κατά δεκτή 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 123 υπέρ κατά αποχές δεκτή 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται εντάξει, εντάξει, ελέγχουμε καλύτερα. Έλεγχος 124. Πέρας. Δεκτή. 125 υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Η ΙΜΚΟ 17 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τραν 11 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 18 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ήμκο 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 126 ε, Πέρα. κατά 126 ελέγχουμε γιατί δεν μπορώ να διακρίνω. Πέρας. Δεκτή. Ήμκο 20 πέρα. Κατά Δεκτή. Ήμκο 21 υπέρ. Παρακαλώ σηκώνετε το χέρι σας. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήμκο 22 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 129 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Εκατόν τριάντα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ήμκο 25 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ήμκο 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Κριστιανά, όταν ξαφνικά σταματάς να ψηφίσεις, δεν ξέρω τι ψηφίζει το ΕΛΚ. Ε, βρες άκρη, βρες την άκρη σου. 132 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ήμκο 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή λίμπε 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή τραν 14 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε την τραν 14 πέρας δεκτή 134 υπέρ κατά ας ελέγξουμε

και ΙΜΚΟ 29 ταυτόσιμες υπέρ, κατά αποχές δεκτές 9 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ, κατά αποχές... Τι ψηφίσατε. 10 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά αποχές 147 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 146 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 32 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή γιούρι συμβαστική 14 υπέρ. Κατά Ας ελέγξουμε. Γιούρι συμβαστική 14. Πέρας. Απορρίπτεται. Λίμπε 20 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 148 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 149 υπέρ. Κατά αποχές. Ας ελέγξουμε την 149. και πέρας απορρίπτεται. Τραν 17 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 150 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή λίμπε 21 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή καλτ 16 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή έμβη 7 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τραν 18 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή 151 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Καλτ 17 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 152 μαζί με την ΙΜΚΟ 34 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Λίμπε 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή, ΙΜΚΟ 35 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 153 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, ΙΜΚΟ 36 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, ΛΥΜΠΗ 23 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 39 19 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 12 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 155 Α, συγγνώμη, 19 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Καλ 20 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Καλ 21 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Καλ 22 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 156 υπέρ, κατά Ας ελέγξουμε την 156. Απορρίπτεται λοιπόν. Κάλτη 23 υπέρ. Κατά. Αποχές αγκρίνεται. Ε, Επιτροπή ε, Υπολογισμού 2 υπέρ. Κατά. Λοιπόν, την υπαριθμό 2 από την Επιτροπή Μπουτζέ, ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τρία Υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να το δούμε και αυτό ηλεκτρονικά. Πέρας απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Λίμπε 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Budgetary 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. NV8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τραν 21 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, κουλτ 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, κουλτ 25 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 158 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τέλος, τελική ψηφοφορία, ονομαστικά, παρακαλώ. Άρχεται. Λοιπόν, ένας ε, παραπάνω από το ΕΛΚ, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται λοιπόν ξεκάθαρα και συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο που είναι η έκθεση που είναι η πρόταση μάλλον για τη θέσπιση του Διαστημικού Προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα. Η συγητής Μασιμιλιάνου Σαλίνη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Να ξεκινήσουμε. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV14 υπέρ. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρειτε MV14. Μπορείτε να τη βρείτε παρακαλώ. NV14 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να το δούμε αυτό. Πέρας. Εγκρίνεται. 1,66 υπέρ, κατά, αποχές, α, για να το δούμε, 1-6-6. Πέρας. Απορρίπτεται. 1,67 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 1,73 υπέρ, Κατά. Α, για να το δούμε ηλεκτρονικά, την 173. Πέρας. Εγκρίνεται. budgetary 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τραν 41 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τραν 57 υπέρ. Κατά. Για να δούμε ηλεκτρονικά. Τραν 57. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δύο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προσθήκη στο συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5-1-8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5-20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5-30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άγκρι 28 υπέρ κατά αποχές 530 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άγκρι 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5.33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5.35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5.46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5.62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5.64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τραν 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τραν 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τραν 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μπατς 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NV2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται NV5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Badge 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Badge 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τραν 12 υπέρ. Κατά αποχές. Για να δούμε ηλεκτρονικά παρακαλώ την επαλήθευση. Τραν 12. Πάλι περισσεύει ένας από το ΕΛΚ. Ο, συγγνώμη, τώρα περισσεύει ένας σοσιαλιστής. Το ΕΛΚ είναι εντάξει. Και οι σοσιαλιστές, εντάξει. Λοιπόν, πέρας ψηφοφορίας για την Τραν 12, απορρίπτεται. Τραν 13 υπέρ, κατά αποχές και αυτήν παρακαλώ ηλεκτρονικά καλύτερα. Τραν 13. Πέρας. Απορρίπτεται. Άγκρι 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 10 υπέρ κατά αποχές. Για να τη δούμε. Τη 10, άγκρι 10. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρασε. Τραν 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. NV8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τραν 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Τραν 24. Επαληθεύουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Ένβι 12 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά παρακαλώ και την ένβι 12. Ηλεκτρονικά. Επαληθεύουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στην ονομαστική τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ξεκάθαρο και θα συγχαρούμε τον εισηγητή μας, τον συνάδελφο Μασιμιλιάνο Σαλίνη. Και μπορούμε τώρα να περάσουμε στην επόμενη ψηφοφορία. Ο κύριος Σιλικιώτης έχει ε, επί της διαδικασίας. Yeah, very short, uh, President. Uh, I want to inform that uh, as a GUE we table... Να σας ενημερώσω ότι ως GUE καταθέσαμε την uh, έκθεση μειοψηφίας για την uh, γνωμοδότηση μειοψηφίας, μειοψηφίας για την έκθεση αυτή. Ωραία, πολύ καλά. Περνάμε στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, ε, εισηγητής ο κύριος Κράσνο Ντέψκι. Θα ξεκινήσουμε. Θα ψηφίσουμε μαζί από την 99 στην 104. Είναι έξι τροπολογίες, ψηφίζουμε μαζί, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα θα περάσουμε. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θα πηγαίνω πιο αργά. Τώρα θέλω να βρείτε την 25, άφετη 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 άφετ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7α υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7α. Ηλεκτρονικά παρακαλώ την συμβιβαστική 7α. Επαληθεύουμε. Καλή ιδέα αυτή να την επαληθεύσουμε. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά. Για να τη δούμε και αυτήν ηλεκτρονικά, γιατί είναι οι συμβιβαστικέ πολύ σημαντικέ. Επαληθεύουμε λοιπόν. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν τώρα στην ΑΦΕΤ 29. ΑΦΕΤ 29 υπέρ. Κατά αποχές και εδώ παρακαλώ ηλεκτρονικά την άφητη 29. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα λοιπόν θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να βρούμε τη συμβαστική 8. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 8α, υπέρ, κατά, αποχές, είναι συμβιβαστική. Η 8α, σας παρακαλώ πολύ, ε, ηλεκτρονικά να επαληθεύσουμε τη συμβιβαστική 8α. 8α, επαναλαμβάνω, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 303. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε την ΑΦΕΤ 38. Ζητήθηκε από τους σοσιαλιστές στην 38 να κάνουμε ονομαστική ψηφοφορία. Είναι 38 άφετ, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εξαιρετικό αποτέλεσμα. Οπότε βλέπετε το σημείο αυτό ε, ταυτιζόμαστε ένας-ένας υπέροχο αποτέλεσμα. 3-3-8 8 υπέρ. 3-3-8 υπέρ. υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να δούμε και την 3, 338 μάλλον ηλεκτρονικά. I close the vote. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 341 υπέρ κατά αποχές και εδώ ηλεκτρονικά παρακαλώ 341 ηλεκτρονικά επαληθεύουμε πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 10 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 357 και 358 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να το δούμε και ηλεκτρονικά. Ωραία, αυτή τη στιγμή είμαστε λοιπόν στις 3.57 και 3.58 τις οποίες ψηφίζουμε μαζί και ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Μαζί, πέρας, απορρίπτεται. 363 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 364 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άφετ 48 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ. Ωραία. Λοιπόν, στην ΑΦΕΤ να πάμε να το δούμε ηλεκτρονικά. Η ΑΦΕΤ 48 παρακαλώ, ηλεκτρονική επαλήθευση. Αγαπητοί φίλοι, έχουν γίνει και λάθη, αλλά ναι, τώρα το δεχόμαστε, κανένα πρόβλημα. Ε, εκτός αν εσείς ε, δεν παίζεται σύμφωνα με τους κανόνες. Συμβιβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, συμβιβαστική 12. Α, συγγνώμη. 368 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Συμβιβαστική 13α. 13α, συμβιβαστική, υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά παρακαλώ να επαληθεύουμε τους συμβιβαστικές γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. 13α λοιπόν πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λοιπόν, συμβιβαστική 14. Μαζί με, με την προφορική τροπολογία και βέβαια θα ήθελα να είμαστε σίγουροι πως στο κατάλογο σας έχετε και την προφορική τροπολογία που έχουμε λάβει από τους πράσινους. Και θα ήθελα να σας πούνε, υπάρχει καμία αντίρρηση στο να έχουμε και την προφορική τροπολογία μαζί. Όχι. Αν έχετε πρόβλημα, σηκωθείτε. Αν έχετε αντίρρηση, παρακαλώ σηκωθείτε. Τέσσερις χρειαζόμαστε. Πέντε σηκώθηκαν. Οπότε, την συμβιβαστική 14, πέντε φτάνουν γιατί σε κάθε επιτροπή χρειάζονται τέσσερις, τέσσερα άτομα. Οπότε ήσασταν και με το παραπάνω αρκετοί. Οπότε πάμε στη συμβιβαστική 14 χωρίς την προφορική τροπολογία, δυστυχώς χωρίς την προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, τροπολογία, εμείς χωρίς αποχή, ε, εγκρίνεται. 16 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4.42 δεύτερο κομμάτι υπέρ κατά Συγγνώμη, πρέπει να το βρείτε. Θα περιμένω. 424 δεύτερο τμήμα μόνο. Είστε έτοιμοι? Είστε όλοι έτοιμοι. Ωραία. 424. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα επαληθεύσουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ. Θα περιμένω. Λοιπόν, είμαστε συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Θα επαληθεύσουμε παρακαλώ, γιατί δεν είναι απόλυτα σαφές. Συμβιβαστική 18. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Αμέσως, γιατί είναι συμβαστική. Είμαστε στη 19 ηλεκτρονικά. Πέρας. Ναι. Εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην... σε τρεις τροπολογίες που είναι οι ίδιες. 450, 451 και 82 ΙΜΚΟ. Υπέρ. Κατά. Για να το επαληθεύσουμε. Είναι τρεις μαζί. Τις ψηφίζουμε και τις τρεις μαζί. Πέρας. Απορρίπτονται. 455 υπέρ. Κατά. Για να το επαληθεύσουμε το την 455. Πέρας. Απορρίπτεται. 456 υπέρ. Κατά. Α, να την ξαναδούμε λοιπόν. 456 πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ξεκάθαρα. 457 υπέρ. Κατά. Παρακαλώ και εδώ ηλεκτρονικά. Δεν είναι ακόμα σαφές για μένα. Πέρας. Απορρίπτεται. Ε, ένα μπιτζέ. Υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Ήμκο 1, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Για να το δούμε. Είμαστε στην 106. Πέρας ψηφοφορίας. 107 υπέρ. Κατά. Και αυτή είναι ηλεκτρονικά παρακαλώ. Η προηγούμενη απερίφθη. 107 πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ήμκο 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2. Μπάτζ. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Του μπάτζ. Πέρας. Απορρίπτεται. Ήμκο 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Budge 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 Ήμκο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αφετ 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά. Για να τη δούμε και ηλεκτρονικά. Είμαστε στην 116. Πέραση της πληροφορία. Εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά. Για να το δούμε. 118. Πέρας. Απορρίπτεται. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 119 υπέρ κατά αποχές για να τη δούμε 119 πέρας απορρίπτεται 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 122 υπέρ έλεγχο ζητείτε για την 121 Ελέγχουμε την 121. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Δίκιο είχατε. Ευχαριστώ. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. 10 τη ΣΥΜΚΟ. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 141 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Για την 141. Πέρες. Απορρίπτεται. 15 της ΣΥΜΚΟ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 153 υπέρ. Κατά, έλεγχος για την 153 παρακαλώ, ελέγχουμε την 153. Πέρας. Απορρίπτεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 11 της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 155 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 της ΕΜΚΟ υπέρ, κατά. Δεν είμαι βέβαιος. 19 της ΕΜΚΟ παρακαλώ. Ας κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ανοίγει η ψηφοφορία. Πέρασε. Μέσα αυτή τη διαφορά βρίσκεται 126 υπέρ 162 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές έλεγχος πέρας ε, απορρίπτεται με 18 αποχές απορρίπτεται λοιπόν 163 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Έλεγχος για την 163 παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. Αυτή τη φορά. Ήμκο 20. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Για τον ΕΜΚΟ 20, παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Οκτώ της Επιτροπής Προπολογισμού υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 171 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23 της ΙΜΚΟ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 173. Υπέρ. Και 174. Από κοινού. Φίλοι μου. Δύο τροπολογίες μαζί. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. Δύο τροπολογίε μαζί πάλι, για 175 και 176 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε αυτές τις δύο παρακαλώ με ηλεκτρονική ψηφοφορία 175 και 176. Πέρασε. Απορρίπτεται. 11 της Επιτροπής υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. 13 αφέτ, υπέρ, κατά. Δεν είναι σαφές. 13 της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, παρακαλώ, ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας της ψηφοφορίας, απορρίφθηκε. 14 της Επιτροπής Εξωτερικών είναι υπέρ. Κατά. Έλεγχος και πάλι παρακαλώ. 14. Ε, δεκατέσσερα της ΑΦΕΤ λοιπόν, πέρασε ψηφοφορίας. Α, αποδεκτό. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 15 παρακαλώ για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων πέρα τη ψηφοφορία τη ηλεκτρονική επαλήθευση. Τώρα εγκρίθηκε. 17 τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. 18 αφέτ υπέρ. Κατά. Έλεγχο. 18 αφέτ. Πέρας. Απορρίπτεται. Τελική πλοίο ε, ψηφοφορία με ονομαστική κλίση, παρακαλώ. Και πέρας ψυχοφορίας; ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια με διαφορά μάλιστα. Και τώρα περνάμε στην επόμενη έκθεση. Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση για τον ΙΤΕΡ και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύνδεξης. Ο εισηγητής μας είναι ο κύριος Μάριαν Μαρινέσκου. Και θα ψηφίσουμε λοιπόν τις τροπολογίες. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Από την πρώτη ξεκινάει. Πέρας ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίφθηκε. 14. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Ας ελέγξουμε και πάλι. Τροπολογία 14. Ε, είναι... Εγκρίνεται με σαφή διαφορά. Δεν χρειάζεται να το ελέγξουμε, αλλά μια και ξεκινήσαμε, να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Πέρασε, πέρασε πάντω. Είναι η τελευταία ψηφοφορία πριν από το διάλειμμα. Σας παρακαλώ κουράγιο να ψηφίζουμε, να σηκώνουμε τα χέρια μας. Πολύ ωραία. 20 δεύτερα να συνταχθούμε, διάλειμμα. Φίλε μου, τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ζητώ συγγνώμη, αλλά φαίνονται αρκετά διαιρεμένα τα πράγματα εδώ πέρα. Πέρας. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 2 υπέρ, κατά. Έλεγχος παρακαλώ για τη συμβαστική 2. Βεβαίως. And I close the vote. της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 Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ. Ελέγχουμε τη συμβαστική 1. Πέρασε. Απορρίφθηκε. 2 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος. Γιατί δύο παρακαλώ ελέγχουμε. Πέρα ψηφορίας. Απορρίφθηκε. Τρία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τέσσερα υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Έλεγχος για την τέσσερα, παρακαλώ. Αλλά έχουμε την τροπολογία υπέρ υπερθμό τέσσερα. Πέρας ψηφοφορίας. Εκρίθηκε. Ένα υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ για την 1. Εξαρτάται από την πολιτική ομάδα φυσικά. Απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος. Η πέντε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίφθηκε έξι υπέρ. Κατά. Με την ίδια πλειοψηφία απορρίφθηκε. έπτα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. οκτώ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. εννέα υπέρ. Κατά. Η ε, 9 ναι, παρακαλώ, να ελέγξουμε την 9. Πέρα ψηφοφορία. Για την 9. 10. Απορρίφθηκε υπέρ. 10. Υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 11. Σε τμήματα. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ. Να ελέγξουμε παρακαλώ το σημείο 2, το δεύτερο τμήμα. Πέρα ψηφορίας. Πέρα ψηφορίας εγκρίνεται 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος, έλεγχος παρακαλώ. Για τη 12. Πέρας ψηφορίας. Τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση προφανώς. Έναξη ψηφοφορίας. Ευχαριστώ πολύ. Εγκρίνεται με σαφή διαφορά. Συγχαρητήρια στον εισηγητή και προχωράμε. Στην επόμενη έκθεση. Έκθεση της Ρεμπέκα Χάρμς. για το πρόγραμμα συνδρομής στον παρακλεισμό του πυρηνικού ηλεκτρικού σταθμού Ιγναλίνα στη Λιθουανία. Η κυρία Ρεμπέκα Χάρπς είναι η συγκεκριά. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Έλεγχος για 13. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Έγκρινεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Έγκρινεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Έγκρινεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Και αυτό έγκρινεται. 53. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 19. Πέρασε. Απορρίπτεται η 1 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Για να είμαστε και σίγουροι. Τροπολογία 2. Πέρα ψηφορίας. Ένας υπεραριθμός ε, από το ΕΛΚΑ. Τροπολογία 2. Μάλιστα. Πέρασε ψηφορία. Ε, εγκρίνεται. Η τρία υπέρ. Κατά. Ας αλλάξουμε και την τρία αν θέλετε. Τροπολογία τρία. Πέρας. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 6 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 25, 26 συγγνώμη και 7 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά αποχές. Ας ελέγξουμε την 9. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Με ονομαστική κλίση τώρα. Η τελική ψηφοφορία. Έναρξη ψηφοφορία. Και πέρασε. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε η έκταση. Συγχαρητήρια στην εισηγητρία. Ε, ε, Group. Οι σοσιαλιστές θα ήθελαν να μας ζητήσουν ε, μία, ένα μικρό διάλειμμα, ένα λεπτό, το οποίο σημαίνει τρία. Αλλά μπορούμε να διακόψουμε και για τρία λεπτά, κανένα πρόβλημα. Ε, Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, ας ε, ξαναρχίσουμε για τα προγράμματα, για το πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ 21-25. Ε, μια πέτρα κουμπούλα νάτρι. Έχουμε τρεις τροπολογίες αν μπλοκ, 58-60-63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Επίσης άλλες τρεις σαν μπλοκ 59, 61, 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 64, 65 υπέρ κατά αποχές δεκτές 66 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται μάλλον, αλλά ελέγχουμε. 66. Έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται, πράγματι. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71-72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 73 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 87 υπέρ κατά αποχές έλεγχος 87 ελέγχουμε πέρας Απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. 89 ελέγχουμε. Πέρας. Και απορρίπτεται. 90 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 91 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 92 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 93 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 94 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 95 υπέρ. Κατά Θέλετε να ελέγξουμε, ας ελέγξουμε λοιπόν την 94. Αμέ με συγχωρείτε, την 95. 95. Έλεγχος. Ψηφίσαμε την 94 πριν 95 λοιπόν. Πέρας. Δεκτή. 96 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε την 96. Πέρας. Απορρίπτεται. Μάλλον. Ναι, 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε την 99. Πέρας. Απορρίπτεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε την 98 έλεγχος. Ένας υπεράριθμος από την ΚΟΕ Εντάξει τώρα, πέρας και απορρίπτεται. 100 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 101 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 102 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 103 υπέρ. Κατά ας ελέγξουμε. 103. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 107 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 129 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 22 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 1 υπέρ. Θέλετε να ελέγξουμε εντάξει. Συμβαστική ένα έλεγχος. Πέρας. Δεκτή. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ. Πρώτο τμήμα. 31 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Ας ελέγξουμε δεύτερο τμήμα της 31. Πέρας και εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ελέγχουμε την 33. Πέρας και απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 39 υπέρ κατά αποχές δεκτή 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή ε, απορρίπτεται συγγνώμη 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή 42 2, 43 μαζί υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται. 45 υπέρ, κατά, ας ελέγξουμε την 45. Πέρας και απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά, ας ελέγξουμε την 46. 46 πέρας. Αποδεκτή 47 υπέρ. Κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε και πάλι. Λυπάμαι αλλά δεν γίνεται αλλιώς. 47 δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Πέρας τώρα. Απορρίπτεται 51 υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε, ας ελέγξουμε. 51. Έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. 1. Ξεχωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα της 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. 48 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 49 και 34 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 50 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 54 υπέρ κατά. Ας ελέγξουμε την 54 καλύτερα. Έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 20 και 21 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Τελική ψηφοφορία με ονομαστική η οποία και αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται σαφώς. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Αγαπητοί φίλοι, Πάμε στην τελική ψηφοφορία πριν από το μεσημεριανό διάλειμμα, αλλά εάν δεν μπορέσουμε να τελειώσουμε μέχρι τις 12.30, όπως ξέρετε, το διάλειμμά μας είναι από τις 12.30. Οι διερμηνείς θα πρέπει να φύγουν στις 12.30 ακριβώς και δεν μπορούμε να ψηφίσουμε χωρίς διερμηνία. Άρα θα σταματήσουμε κάποια στιγμή και το υπόλοιπο θα συνεχιστεί, η ψηφοφορία δηλαδή, στις 2.30 και τότε θα ολοκληρώσουμε την ψηφοφορία. Τώρα θα ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα και θα σταματήσουμε στις 12.30 ακριβώς και θα ολοκληρώσουμε από τις 2.30 και μετά. Εντάξει, είμαστε σύμφωνοι. Ωραία. Ας προχωρήσουμε. Σχέδιο γνωμοδότησης του συναδέλφου Ζωάου Φερέιρα. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής. Γνωμοδοτούμε και για τα δύο ταμεία. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 1. Ε, ας ελέγξουμε. Ας ελέγξουμε την 113. Ηλεκτρονικά. Συμβιβαστική, μάλλον τη συμβαστική 1 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας απορρίπτεται. 114 υπέρ, κατά, αποχές δέκτη 22 υπέρ, κατά, ας ελέγξουμε την 22, πέρας, απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 115 υπέρ κατά ας ελέγξουμε την 115 πέρας απορρίπτεται 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή 117 υπέρ κατά αποχές δεκτή 22 υπέρ με συγχωρείτε 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε 26 Απορρίπτεται. 119 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 120 υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε. Είκοσι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 121 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε. Την 123 ελέγχουμε. Πέρας απορρίπτεται. 124 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, δεκτή. 125 υπέρ, κατά. Έλεγχος παρακαλώ. 125 ελέγχουμε. Πέρας. απορρίπτεται. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε καλύτερα. Ας ελέγξουμε. Πολύ απήχαν. Πέρας. Και απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε την 30. 30 ελέγχουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 129 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. 129 ελέγχουμε. Πέρας. Δεκτή. 130 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. 130. Έλεγχος. Πέρας. Και απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 132 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή 133 υπέρ κατά αποχές δεκτή 134 υπέρ κατά αποχές δεκτή 135 υπέρ κατά αποχές Ας ελέγξουμε. 135. 135. πέρας δεκτή 136 υπέρ κατά αποχές δεκτή 137 υπέρ κατά πρέπει να ελέγξουμε βεβαίως 137 Πέρας. Απορρίπτεται. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η επόμενη αποσύρεται. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ελέγχουμε την 35. Πέρας. Και απορρίπτεται. 141 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. 140 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε την 140. 140 έλεγχος. Δεν σηκώνετε το χέρι όπως θα έπρεπε. Τι να σας κάνω. Πέρας. Αποδεκτή. Σαφέστατα. 143. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 144 υπέρ κατά αποχές δεκτή 36. έξι. Αλλά αγαπητοί φίλοι, στην περίπτωση της 142 θα πρέπει επίσης να ψηφιστεί γιατί υπερψηφίσαμε την 140 και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ψηφίσουμε την 142 ώρα πριν την 36. Πάμε τρεις πίσω και ψηφίζουμε την 142. 142. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 142. Πέρας. Δεκτή. Τώρα. Πάμε απευθείας στην 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 145 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Στην 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές για να το δούμε ηλεκτρονικά. Για την 147 παρακαλώ. Εγκρίνεται. Η 147 εγκρίνεται. 149 Συγγνώμη. 148 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 149 υπέρ. Κατά. Για να το δούμε ηλεκτρονικά στην 149. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικά παρακαλώ και εδώ. Πέρας ψηφοφορίας. απορρίπτεται. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονικά παρακαλώ. Για την 152 ηλεκτρονική επαλήθευση πέρας ψηφοφορίας Απορρίπτεται. 100, ε, η 40 υπέρ. Κατά. Την τροπολογία 40 υπέρ υπαλληθεύουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Με την ίδια ψήφη πλειοψηφία 140, ε, συγγνώμη, η 42 υπέρ. Κατά. Λοιπόν, συγγνώμη, στην 154 είμαστε, ηλεκτρονικά. 154, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 155, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 42, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Για να τη δούμε ηλεκτρονικά τη 43. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ. Κατά. Για να το δούμε ηλεκτρονικά, 45 ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 159 υπέρ κατά ηλεκτρονικά παρακαλώ την 159 πέρας απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 160 υπέρ κατά ηλεκτρονικά παρακαλώ την 160 160 πέρας ένας παραπάνω από την κούε ήσασταν εντάξει απορρίπτεται 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά πρέπει να τη δούμε ηλεκτρονικά τη 48 θέλω να τη δούμε ηλεκτρονικά πέρας απορρίπτεται 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 163 υπέρ κατά ηλεκτρονικά παρακαλώ την 163 163 πέρας απορρίπτεται 164 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 167 υπέρ κατά για να δούμε ηλεκτρονικά 167 167 πέρας. Απορρίπτεται 169 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά παρακαλώ, την 169. 169. Πέρας. Απορρίπτεται. 51 D υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 118 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά παρακαλώ την 156. 156 παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2. Εδώ θα ήθελα ηλεκτρονικά παρακαλώ. Συμβιβαστική 2. Πέρας. Εγκρίνεται με ξεκάθαρη πλειοψηφία. 190 και 193 μαζί, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και οι δύο απορρίπτονται. Περνάμε τώρα στην 198. 198. Υπέρ. Κατά. Για να τη δούμε ηλεκτρονικά. 198. Πέρας. Απορρίπτεται. 199 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 200 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 201 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 202 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 203 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 204 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 157 υπέρ α, με συγχωρείτε Έχουμε εγκρίνει τη 204, τώρα πάμε στη 206 κατευθείαν. Συνάδελφοι, στη 206 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 207 υπέρ. Κατά. Για να δούμε ηλεκτρονικά με τη 207 τι γίνεται. 207. Πέρας ψηφοφορίας. 207. Εγκρίνεται. «208 υπέρ». Κατά. Απορρίπτεται. 209 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 210 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 211 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 59 του κυρίου Φερέιρα αποσύρεται. Εξ όσων γνωρίζουμε. Απορρίπτεται. Η, με συγχωρείτε. η 58. Η 58 αποσύρεται, την 59 ψηφίζουμε. Για, εξηγήστε μας, κύριε Φερέιρα. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε σφάλμα στον κατάλογο ψηφοφοριών. Δεν ψηφίζουμε την 59. Την 58 πρέπει να την ψηφίσουμε. Είναι λάθος ο κατάλογος. Γιατί η τροπολογία 201 έχει αντικαταστήσει την 59 και όχι την 58. Οπότε θα ψηφίσουμε την 58 και όχι την 59. Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι που δεν είδαμε προηγουμένως το σφάλμα αυτό. Ναι, εντάξει, είναι ο εισηγητής μας, οπότε αυτό που λέτε εσείς αυτό ισχύει. Περνάμε τώρα στην 59 που δεν θα ψηφιστεί και την αφήνουμε στην άκρη και αυτή τη στιγμή θα ψηφίσουμε την 58. Υπέρ. Κύριε Πρόεδρε, την 58 δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε γιατί δεν είναι στον κατάλογο για την 58 αναβάλλεται την ψηφοφορία μέχρι μετά το διάλειμμα και την ψηφίζουμε τότε. Okay. Uh, because, uh, we probably cannot... Ναι, έτσι κι αλλιώς δεν θα τελειώσουμε. Αν δεν υπάρχει όμως άλλη δυνατότητα, μπορούμε να σταματήσουμε τις ψηφοφορίες και να πούμε πριν την ονομαστική θα την ψηφίσουμε. Ωραία. Αφήνουμε την 59 γιατί δεν θα την ψηφίσουμε και την 58 θα την ψηφίσουμε πριν ξεκινήσω την τελική ονομαστική ψηφοφορία. Οπότε σίγουρα μετά τη μεσημεριανή διακοπή, αγαπητοί φίλοι. Σίγουρα μετά τη μεσημεριανή διακοπή και γι' αυτό σκεφτείτε την 58 τι θα την, πώς θα την ψηφίσετε. Ακριβώς λοιπόν πριν την τελική ονομαστική ψηφοφορία. Τώρα να περάσουμε στην 59, την οποία δεν ψηφίζουμε, να την αφήσουμε και να περάσουμε στη 212. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Τη συμβαστική 3 ηλεκτρονικά πέρας. Απορρίπτεται. Οπότε. Βλέπουμε τη 213. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 214 και 60 μαζί υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 69, 61 με συγχωρείτε D υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 215 και 216 μαζί υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 217 υπέρ κατά ηλεκτρονικά παρακαλώ. 217 Πέρας. Απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 218 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να τη δούμε ηλεκτρονικά. 218. Παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 63D in favor. Λοιπόν, περνάμε μετά στην 223D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, συγγνώμη, αυτή ήταν η η 63. Τώρα 220 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 222 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 221 υπέρ κατά αποχές. Τη 221 παρακαλώ επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 223 υπέρ. Κάτα. Επαληθεύουμε τη 223 παρακαλώ. Ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. Δύο τροπολογίες, 224 και η 64 μαζί, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 65D υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 225 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 227 υπέρ κατά Είμαστε στη 227. Για να τη δούμε. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 228. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 229. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 230 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.31 υπέρ. Κατά. Για να τη δούμε ηλεκτρονικά. 2.31. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.32 υπέρ. Κατά. Αποχές και πάλι ηλεκτρονικά παρακαλώ. Είμαστε στη 2.32. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 233 υπέρ. Κατά. Και άλλη μια φορά λοιπόν ηλεκτρονικά παρακαλώ. Τη 233 παρακαλώ να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. 67D υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα περνάμε στην τροπολογία 280, δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 281, δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 282 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 283 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά, παρακαλώ τη 283. Για να τη δούμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Αγαπητοί φίλοι, έχουμε τα παραρτήματα. Η πρότασή μου είναι να σταματήσουμε εδώ, γιατί έχουμε ένα-δύο λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, και μετά μην ξεχάσετε πως επιπλέον θα ψηφίσουμε και αν δεν κάνω λάθος, την τροπολογία υπαριθμών 58 πριν την τελική ψηφοφορία. Και θα ξεκινήσουμε με το παράρτημα 2 πίνακας πρώτος, μόλις γυρίσουμε από τη μεσημερινή διακοπή στις 2.30.